Αγαπητοί συνάδελφοι, meeting... μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε αντιρρήσει στο σχέδιο ημερησίας διατάξεως εγκρίνεται ανευτροποποίησεων και τώρα πρέπει να ξεκινήσω με τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Πρώτη ανακοίνωση. Σχετίζεται με διορθωτικό στον αυτόν τον κανονισμό 536 του 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές ετρικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και την ε, ανάκληση οδηγίας κλπ. Εδώ έχει εντοπιστεί ένα σφάλμα στον κανονισμό 536 όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σχετική θέση σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου του 2014. Το σφάλμα αφορά ασυνέπεια του κειμένου των διατάξεων του άρθρου 8.5, 19.3 και 23.5 που είναι σχεδόν ε, ταυτόσιμα αυτά τα τρία άρθρα στη διατύπωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζητήθηκε από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσει με την προτινόμενη διόρθωση του σφάλματος. Λοιπόν, ένα διορθωτικό προς έγκριση έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με το άρθρο 231. Η αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει το σχέδιο διορθωτικού κειμένου και θα το υποβάλει στο Κοινοβούλιο αν θεωρεί ότι πράγματι έχει διαπραχθεί ένα σφάλμα το οποίο μπορεί να διορθωθεί με τον προτινόμενο τρόπο. Το διορθωτικό απεστάλλει σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος την Τετάρτη. Αν δεν ε, υπάρξουν ε, αντιρρήσει μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδριά της Επιτροπής, το διορθωτικό θα θεωρηθεί εγκεκριμένο και θα υποβληθεί δεόντως το Κοινοβούλιο προς ανακοίνωση στην, ε, στη σύνοδο της, ε, στην πρώτη σύνοδο του Οκτωβρίου. δεύτερη ανακοίνωση αφορά την έκθεση ε, ΑΦΚΟ για την αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού. Προτείνει η Επιτροπή ΑΦΚΟ γενική αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου που θα τεθεί σε ισχύ ε, εσωτερικός κανονισμός στη Σύνοδο του 2017 του Ιανουαρίου. Η αναθεώρηση αφορά διάφορα θέματα σημαντικά που αφορούν τις εργασίες Επιτροπής Περιβάλλοντος, πρωτίστως δια, ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά νομοθετικά θέματα. Το χρονοδιάγραμμα της ΑΦΚΟ είναι πολύ φορτωμένο και έχει σχεδιαστεί ψηφοφορία 8 Νοεμβρίου για να μπορέσουμε να δώσουμε στην, ε, τις απόψεις της όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, οι συντονιστές αποφάσισαν να καθορίσουν προθεσμία για τροπολογίε στα αγγλικά μόνο όσον αφορά το σχέδιο εκθέσεως της ΑΦΚΟ για την 5η-6 Οκτωβρίου το, μεσ... Οκτωβρίου το μεσημέρι. Η ψηφορία θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου και οι τροπολογίες που θα υιοθετηθούν θα συμπεριληφθούν στην ε, γνωμοδότηση. Έχουμε ερμηνεία 21 γλώσσες και ε, Έχετε επίσης και τη, θα έχετε και τις σημειώσεις για τη συνεδρίαση ηλεκτρονικά. Πάμε τώρα στην ψηφοφορία. Πρώτη ψηφοφορία όσον αφορά τα, τα, τα λύπη, τα, τα τάνς Και αν είστε έτοιμοι θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 54, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τροπολογία 66 ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 68 υπέρ. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να ψηφίσουμε την 69, τροπολογία 69, 68 καταπίπτει. Τροπολογία 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 71 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται τώρα συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα την τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27, υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική μονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Έγκρινατε. Συγχαρητήρια. Το επόμενο σημείο. Στατηγική αεροπορική για την Ευρώπη. Ξεκινάμε με τη συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας με παρουσίαση της γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος η Επιτροπή Μεταφορών όσον αφορά εφοδιαστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολυτροπικές μεταφορές τους ε, νέους διαδρόμους καλό όλα τα μέλη που δεν ενδιαφέρονται στη συζήτηση που θα διεξαχθεί να, να αποχωρήσουν σύντομα από την αίθουσα, παρακαλώ, και έτσι θα μπορέσει ο κ. Τσόφολη, ο εισηγητής μας, να παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε και παρακαλώ τις συζητήσεις σας αν έχετε την καλοσύνη να τις κάνετε έξω. Κύριε Τσόφολη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή των Μεταφορών πρέπει να γνωμοτήσει επί πρωτοβουλίας που αφορά ε, την, εφοδιαστική όσον αφορά τα συστήματα, τα πολυτροπικά των μεταφορών στους διαδρόμους ΤΕΝΤΗ. Μιλάμε για έναν τομέα στρατηγικής σημασίας, την αλυσίδα αυτή της ε, οργάνωση που αφορά το 13% του ΑΕΠ στην ε, Ευρώπη, 15% του κόστους των ε, καταργασμένων προϊόντων, ψυχασμένων προϊόντων που εξαρτώνται από την όλη εφοδιαστική αλυσίδα. Το αίτημα που υπευλήθη, υπευλήθη στην Επιτροπή να εκπονήσει μια νέα στρατηγική όσον αφορά την εφοδιαστική για τα εμπορεύματα μέχρι το 2017, λαμβάνοντα υπόψη και τις μεγάλες αλλαγές και την κρίση που ζούμε και τους πρόσφυγες που έχουν συνέπειες όλα αυτά και για τη μεταφορά ε, των εμπορευμάτων, το Brexit και αφορά και το περιβάλλον, οι διάφορα διάφορα που καταβάλλονται στο COP21 Παρίσι αναλάβαμε υποχρέωση να μειώσουμε κατά 40% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τομέας των, μεταφορά, των μεταφορών εκπέμπει περίπου τον τέταρτο συνολικά εκπομπωμένων μεταφορών και τα δύο τρίτα των εκπομπών αυτών εξαρτώνται από τις οδικές μεταφορές. Είναι προφανές λοιπόν ότι το κρίσιμο σημείο είναι η βιωσιμότητα των μεταφορών, κυρίως των οδικών μεταφορών, που χρησιμοποιείται περισσότερο διότι κοστίζει λιγότερο η οδική μεταφορά όσον αφορά ε, χρόνο και τιμές και κόστος. Πέρα και από τις συνήθειες βέβαια. Ε, θα πρέπει να αλλάξουν γενικά οι συμπεριφορές και οι νοτροπίες. Όσον αφορά τις συμπεριφορές και την νοτροπία, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη διάδοση της στρατηγικής just in time, όταν φτάνουν τελευταία στιγμή, ακριβώς την ώρα τους τα εμπορεύματα. Μειώνουμε ε, στον ελάχιστο αριθμό της αποθήκευση, αυξάνοντας τα οχήματα που κινούνται, διότι η κινητικότητα των εμπορευμάτων ε, εξαρτάται άμεσα από τη ζήτηση έχουμε διεξαγάγει μια συζήτηση για πόλεις. Μιλάμε για μια κυκλική οικονομία και είναι σημαντικό αυτό. Μιλάμε για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξη με την κυκλική οικονομία. Τι σημαίνει κυκλική οικονομία. Σημαίνει απόβλητα και υλικά τα οποία δεν είναι προβλήματα αλλά είναι πλέον πηγές, πόροι. Δεν είναι απορρίμματα, είναι πηγές. Έχουμε πρώτες ύλες, δευτερογενείς ύλες, υποπροϊόντα, ε, υλικά προς νέα χρήση, προς ανακύκλωση, να προς αναγέννηση είναι το Είναι λοιπόν εμπορεύματα τα οποία κυκλοφορούν και που σήμερα δεν έχουν ενταχθεί στην, στο εφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς εμπορευμάτων. Εμείς ασχολούμαστε με το θέμα το εφοδιαστικό διανομής, αλλά έχουμε και αυτή την καινοτομία ε, που αφορά την αντίστροφη εφοδιαστική, δηλαδή πώς μεταφέρουμε ε, αυτά τα υλικά ε, που ανέφερα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, τα ανακυκλώσουμε κλπ. κρίσιμα σημεία λοιπόν είναι δύο. Η μείωση των εκπομπών ε, των αερίων του θερμοκηπίου, της ρήπανσης ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά και της ηχητικής ρήπανσης, της χορύπανσης. Ε, άλλο ένα κρίσιμο σημείο αυτό. Δηλαδή από την εφοδιαστική το 80% ε, ε, των κατοίκων της Ευρώπης κατοικούν σε αστικά κέντρα. Οπότε ε, έχουμε την κρίση του τελευταίου κομματιού της διαδρομής. Ξέρουμε τι σημαίνει η συμφόρηση που προκαλείται. Τι σημασία έχει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα να φτάσουν στα αστικά κέντρα τα εμπορεύματα. Μιλώντας για την εφοδιαστική σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να μιλήσουμε για σχεδιασμό. Θα πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε αν θέλετε σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται ένα σχεδιασμός ε, αλλαγή σχεδιασμού κατά 360 μοίρες, ολοκλήρωση ε, των πολιτικών των κρατών μέλων, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και, τον, και του δημόσιου τομέα των διαφόρων ιδιωτικών φορέων. Χρειάζεται τα μέσα μεταφοράς να είναι ολοκληρωμένα, να θέλουμε να υπάρχει συνδυασμός μεταξύ τους, εσωτερική ναυσιπλοή, οδικές μεταφορές, υδρομικές, ε, ποτάμιες μεταφορές, θαλάσσιες, εναέριες μεταφορές. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τι πηγέ, ε, τα χρήματα, τι πρώτε ύλε κλπ. Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική που απαιτεί ένα σχεδιασμό, ξεκινώντα από μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα στοιχεία και τι πληροφορίε. Πρέπει να μοιράζονται οι πληροφορίε. Χρειάζεται μια ε, πρόσβαση στι ροέ και στα στοιχεία, άρα είναι στατική σημασία να γίνουν επενδύσει όσον αφορά την ψηφιοποίηση του τομέα ε, χρειάζεται μια επένδυση που θα πρέπει να φτάσει και μέχρι τα τερματικά, μέχρι, τις, μέχρι τα άκρα. Όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα, αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν οι μικρές επιχειρήσεις το 90% ε, των παραγωγικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και θα πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις οι μικρές να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ε, και να ενδιαφερθούν για τις αλλαγές. Αυτό αν θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι και ζήτημα ενημέρωσης, εκπαίδευσης του προσωπικού, κατάρτισης. Ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει δυνατότητα νέων θέσεων απασχόλησης ποιοτικών θέσεων απασχόλησης στον τομέα. Πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται, πώ αντιμετωπίζει το κοινωνικό ε, dumping, όπως είναι αυτοσχέδιο οδηγή ε, φορτηγών με 500, 500 ευρώ πληρώνονται αυτοί οι οδηγοί, πολύ χαμηλή, χαμηλή αμοιβή, ε, είναι ε, ερασιτέχνες οδηγοί αυτοί, δημιουργούνται ατυχήματα και προβλήματα λόγω αυτής της ε, κίνησης. Χρειάζεται στρατηγική ολοκληρωμένη προσέγγιση να ληφθούν υπόψη όλες οι πτυχές ε, του τομέα. Τώρα πιο συγκεκριμένα, λέω κλείνοντας, αν ο στόχος είναι αυτός που θέλουμε, δηλαδή να μεταφέρουμε εμπορεύματα και να υπάρχει συμμετοχή τους στον σιδηρόδρομο των δικών μεταφορών, χρειάζεται έρευνα, χρειάζεται καινοτομία, τεχνολογική καινοτομία, χρειαζόμαστε τρένα πιο μακρά, με πιο πολλά βαγόνια, πιο γρήγορα, μεγαλύτερα δυνατότητα, μεγαλύτερες δυνατότητες ε, μεταφοράς φορτίων, χρειάζεται και συντήρηση. Ε, δεν χρειάζεται μόνο νέε επενδύσει στου ιδεοδρόμου, χρειάζεται και η σωστή ε, συντήρηση των υφισταμένων σειρμών. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Μιλήσαμε για τους στρατηγικούς διαδρόμους που πετούνται των τέντη των διαευρωπαϊκών δικτύων. Αυτοί οι διάδρομοι δεν θα πρέπει να παραμείνουν ε, απομονωμένες διαδρομές. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό πράσινο ολοκληρωμένο δίκτυο ε, με διασυνδέσεις όπως και δευτερεύουσες διασυνδέσεις ε, που πρέπει να συμμετέχουν στο δίκτυο. Ε, αυτή είναι η πολιτική, θα πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να γίνουν επιλογές. Αυτά είναι κάτι που πειράζει το κόστος. Είδαμε πως οι τιμές καθορίζονται από την επιλογή των μέσων μεταφοράς. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα ε, τελών, τιμολόγησης, διοδίων, κινήτρων, αντικινήτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή ότι εκείνο που χρησιμοποιεί πληρώνει, εκείνο που ρηπαίνει πληρώνει. Ε, να εφαρμόζονται, δεν θα πρέπει να παραμένουν σύνθημα. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα, κυρίω για τι αστικέ περιοχέ, ε, τη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων. Να υπάρχουν υποδομέ για εναλλακτικά καύσιμα. Να μειωθεί η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στι περιοχέ τι αστικέ. Ε, σε αυτό το τομέα αληθεύει ότι οι πολιτικέ είναι στα χέρια τη τοπική αυτοδιοίκηση αλλά η Ευρώπη πέρα από να ευνοεί την ανταλλαγή των καλών πρακτικών μέσω του συμφώνου των δημάρχων που θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δήμων θα πρέπει να έχουμε συμμάχους και τους πολίτες και τους δημάρχους, τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδίκησης που κάθε μέρα ζουν με τις κοινότητες τους τις δυσκολίες, τις συγκεκριμένες δυσκολίες, το πρόβλημα των ε, απορριμμάτων ε, και της ρήπανσης ε, των μεταφορών το ζουν καθημερινά οι άνθρωποι. Αν θέλουμε να ξανασυνδεθεί η Ευρώπη με τους πολίτες θα πρέπει να διαφερθούμε για αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, να ασχοληθούμε με τα θέματα μετά που φτάνουν στο τέλος την καθημερινότητα της ζωής των πολιτών επηρεάζουν την καθημερινότητα της ζωής των πολιτών μας των ανθρώπων μας Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα σημεία τα οποία εξετάζονται στην έκθεση της πρωτοβουλίας. Εγώ υπογράμμισα τις πτυχές που αφορούν περισσότερο τη βιωσιμότητα, την αηφορία στον αφορά το περιβάλλον. Ε, σαφώς η γνωμοδότηση είναι ατελής, χρειάζεται χρόνος για την ολοκλώρησή της. Μέχρι 11 Οκτωβρίου έχουμε προθεσμία για τις ε, τροπολογίες και περιμένω συνεργασία με τους συναδέλφους και συνεισφορά από πλευράς όλων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο εισηγητή και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων, να ακούσουμε τους κοιόδης εισηγητέ. Ο κύριος Νταντέν έχει το λόγο. Κύριε Νταντέν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. αντικαθιστώ τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ που ζητάει συγγνώμη και τον κύριο Καντάν δηλαδή και εγώ θα σας παρουσιάσω την παρέμβασή του. Αγαπητοί συναδελφοί, ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρότασή του που θεωρώ ότι αποτελεί μια καλή βάση εργασίας. Συμφωνώ με τα διάφορα σημεία που υπογράμμισε ο εισηγητής, κυρίως όσον αφορά την ε, στρατηγική μας για να απαλλαγούμε από τον άνθρακα στις μεταφορές. Είναι για το περιβάλλον και βασίζεται και στη Συμφωνία των Παρισίων. Οι πολυτροπικές μεταφορές επίσης θα βοηθήσουν να μειώσουμε την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον ε, κυρίως μεταφερθούν οι μεταφορές από τις οδικές στις σιδηροδρομικές, κυρίως μιλάω εδώ για τις εμπορικές μεταφορές. Δύο θέματα πιστεύω ότι έχουν προτεραιότητα εδώ. Το ένα είναι να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ο ηλεκτρισμός στις μεταφορές 94% των εμπορικών μεταφορών στην Ευρώπη σήμερα εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη ανεξαρτησία μας. Οι ηλεκτρικές μεταφορές επιτρέπουν λιγότερο αποτύπωμα άνθρακα και επιπλέον στις πόλεις δίνουν καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερο κόστος ανά χιλιόμετρο. Δεύτερον, πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε, να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε δεδομένα, να υπάρξει μια ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής. Γι' αυτό θα ήθελα να αναπτυχθεί μία μέθοδος λογιστική ουσιαστικά που να καταγράφει την κατάσταση όσον αφορά τον άνθρακα και τρύπαση της ατμόσφαιρας στις εμπορικές μεταφορές. Θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό συμβασμό για το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντόρμαν τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την επεξεργασία του σημαντικού αυτού θέματος μιλούμε για τις μεταφορές και για κτηριακές υποδομές που παράγουν διοξείδιο του άνθρακος. Μην δυσμονούμε ότι καμιά φορά κινητοποιούνται κιόλα τα μεγάλα οχήματα. και τα τρένα που θα παραλάβουν το εμπόρευμα από τα φορτηγά αυτοκίνητα πρέπει να φτάσουν στην ώρα τους. Φανταστείτε για τα τρένα που φεύγουν προς τις σκανδιναβικές χώρες. Θα είναι ευκολότερο λοιπόν να χρησιμοποιηθούν φορτηγά μεγάλης χωρητικότητας. Το άλλο θέμα είναι η ασφάλεια στους δρόμους μας με αυτά τα μεγάλα βαριάς χρήσης φορτηγά αυτοκίνητα πώς μπορούμε να τα κάνουμε ασφαλέστερα τα οχήματα αυτά. Διότι έχουμε δει ότι η κατανάλωση υνοπνεύματος και μεταξύ των επαγγελματιών οδηγών αυξάνεται και θα χρειαστεί θα χρειαστεί να φοδιάσουμε τα οχήματα αυτά με μηχανήματα, με αισθητήρε που θα ε, αντιλαμβάνονται εάν έχει ε, καταναλώσει ενόπλο οδηγό και θα αρνούνται να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Εάν η εφοδιαστική λειτουργήσει καλά, η συνεργασία με το, με το σιδηρόδρομο είναι πάρα πολύ σημαντική. Αναμένω με ενδιαφέρον την περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάτιν Μάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο εισηγητής στην αρχή της τοποθετήσεώς του, οι μεταφορές λόγω των μεταφορών εκλείονται δηλαδή περίπου τα 25% των αερίων θερμοκηπίου. Αν θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε αποτελέσματα, πρέπει να μπορέσουμε να μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές καυσαερίων των ε, μεταφορών. Χρειάζεται ανάληψη δράσης στην πράξη και αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγή συνηθιών, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω. Θα γίνουν αλλαγέ, και θα χρειαστεί να γίνουν αλλαγέ. Θα πρέπει να έχουν ωστόσο και την ελευθερία οι χώρες μέλη να πειραματιστούν με τρόπους μείωσης των αερίων θερμοκηπίου θα υπάρξουν ίσως και σφάλματα στην πορεία. Χρειαζόμαστε μια βαθιά αλλαγή στις μεταφορές. Και δεν μιλούμε μόνο για κινητά τηλέφωνα, FE, κινητά τηλέφωνα και ούτω καθεξής. χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις και εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και από την υπόλοιπη κοινωνία. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει λόγο, ρόλο πρωτοπόρο. Μιλώ εδώ τώρα και για την έδρα του Κοινοβουλίου, για τις ε, δύο, την διπλή έδρα του Κοινοβουλίου, η οποία στην ουσία συνεπάγεται μια εντελώς περιττή κινητικότητα που οδηγεί εν τέλει στην έκκληση ε, σημαντικών ποσοτήτων αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Εδώ χρειάζεται να αλλάξουν νοοτροπία οι χώρε μέλη. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να αυξηθεί και η αποδοτικότητα στη χρήση της ενέργειας μεταφορές και προσώπων και αγαθών. Ρίξτε μια ματιά στην ε, λεωφόρο Μπελιάρ περνάει από εδώ κοντά και θα δείτε ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα κινούνται με ένα μόνο επιβάτη, τον οδηγό. Χρειάζεται να στραφούν στα δημόσια μέσα μεταφοράς που εκλείουν πολύ λιγότερα αναλογικά καυσαέρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γιατί ξέρετε το κείμενό του και με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω την περαιτέρω εξέλιξη. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you, Chair. Um, has asked me just to... Κυρία Νόλε, ευχαριστώ πολύ. Πολλά είναι τα θέματα τα οποία αναφέρονται. Χαιρόμαστε για την προσπάθεια της Επιτροπής ε, όσον αφορά τις προδιαγραφές για τα εμπορικά οχήματα και τα όρια διοξιδίου του άνθρακος, αλλά νομίζουμε ότι μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μακριά. Πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει βλέπουν τα εμπορικά οχήματα σαν μεγάλο πρόβλημα και υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα όσον αφορά τα όρια του διοξιδίου του άνθρακα. Αλλιώς θα πρέπει και εμείς περισσότερο να ερευνήσουμε το θέμα του Dieselgate. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας αφορά και όμως 25% της χρήσης καυσίμων στους δρόμους οφείλεται σε 5% των οχημάτων. Δεν υπάρχει πρόοδος πάντως μέχρι τώρα και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πολλά θέματα αναφέρονται όντως για σταθμούς όπου μπορεί κανείς το ηλεκτρικό του όχημα να το φορτίσει που δεν υπάρχουν ε, προς το παρόν και νομίζω ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στα τέντη για να βοηθηθούν οι οδηγοί. Η σκιώδη συζητήτριά μας τονίζει ότι υπάρχουν οικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων επειδή ερμηνεύεται πάρα πολύ αυστηρά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αλλά η συλλογικότητα βοηθάει και τον κόσμο και τις επιχειρήσεις σε ανάπτυξη. Αλλιώς οι προοπτικές καταστρέφονται για να έχουμε ένα καλό κοινωνικό και οικονομικό μέλλον. Η Ιρλανδία από όπου προέρχομαι εγώ έχει πρόσφατα περάσει από οικονομικές και δημοσιονομικές εμπειρίες και είναι μια χώρα η οποία έχει σημαντικά παραδείγματα όσον αφορά τους σιδηροδρόμους. Ελπίζω να συνεχίσει επιτυχία στο δυτικό τμήμα με τους δρομοδρόμους. Έχω υποβάλει σχετικά τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Από το e η κυρία Χέντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον συνάδελφο για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που παρουσίασε. Ε, αναγνωρίζω τις θετικές πτυχές που περιλαμβάνονται ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τάχιστα τις διάφορες προκλήσεις του τομέα το πολυτροπικού δικτύου μεταφορών. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα για να έχουμε καλύτερη βιωσιμότητα. Κυρίως πρέπει να γίνουν προσπάθειες για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της COP21. Θα ήθελα όμως να επιμείνω επί κάποιων στοιχείων που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής όπως το ότι πρέπει να αυξήσουμε την ενεργητική απόδειξη στον τομέα, στο διατροπικό, στις τροπικές μεταφορές, όσον αφορά την εφοδιαστική. Και κυρίως το δικές μεταφορές, η Λευκή Βίβλος για τη μεταφορά του 2011 καθορίζει σαφή κριτήρια, πολύ σαφή κριτήρια όσον αφορά τις διαδρομέ πάνω από 300 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Λευκή Βίβλο, το 30% των μεταφορών των εμπορευμάτων επί των, επί οδών θα πρέπει να, να πάει με άλλου τρόπου όπως ε, μέσω ναυσιπλοεία ή συνδρομικό μεταφορό μέχρι το 2030 και το 2050 θα πρέπει αυτό το ποσοστό να γίνει 50%. Θα ήθελα να υπογραμμίσω άλλε ε, δύο πτυχέ που θεωρώ ότι είναι σημαντικέ. Χρειάζεται να υπογραμμίσουμε λοιπόν σε αυτό σε αυτό το έγγραφο την ανάγκη που υπάρχει, απόλυτη ανάγκη, να είναι δεσμευτικές οι περιβαλλοντικές επιταγές όσον αφορά την αδειοδότηση των διαφόρων έργων υποδομών που, ασχολούνται με το θέμα της εφοδιαστικής. Θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει το δημόσιο περισσότερο το, στις αποφάσεις και το κοινό να συμμετέχει στις αποφάσεις που θα, για έργα που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες διάφορες κοινότητες. Τέλος, πιστεύω ότι πέρα από την αύξηση διαφάνειας των διαδικασιών λήψης αποφάσεως για να χρησιμοποιούνται σωστά τα χρήματα της Ένωσης και των κρατών μελών πρέπει να χρησιμοποιούνται λογικά. Χρειάζεται εξυγχρονισμό των δικτύων και των κόμβων. Χρειάζεται απ' την άλλη και επανεξέταση των υπερβολικά μεγάλων έργων. Θέλω να το υπογραμμίσω, που βασίζονται πολύ συχνά επί πολύ αισιόδοξων προβλέψεων όσον αφορά τι ροέ τη κυκλοφορία που δεν είναι πολύ ρεαλιστικέ. και δεν σέβονται αυτά τα προγράμματα την πραγματικότητα. Και τελικά αυτά τα έργα μπορεί να μην είναι βιώσιμα οικονομικά και να είναι και επικίνδυνα τα έργα αυτά για το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Πίτερ Ντεμέιρο, ονομάζομαι από την Γενική Διεύθυνση MOVE. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον όλε τι παρεμβάσει των εισηγητή, του και όλες εισηγητές, του βουλευτέ για τι απόψει του όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειε όσον αφορά τι προτάσει, Επιβεβαιώνω όμω ότι για τι περισσότερε δράσει και προτάσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει τι δικέ τη προτάσει. Πρόσφατα ε, ετοιμάσαμε και μία ανακοίνωση για την κινητικότητα χαμηλού άνθρακα. Η γνωμοδότησή σας ε, λοιπόν θα πάει στην Επιτροπή Τραν και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην Τραν και με ιδιαίτερη χαρά θα συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σας ε, για αυτήν την τόσο σημαντική πρόκληση. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Και τώρα για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα μετά από τη συζήτηση αυτή ο εισηγητής μας, ο κύριος Τσαφόλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ να επενθυμίσω την προθεσμία της 11 η Οκτωβρίου που είναι αρκετά κοντά για την υποβολή των τροπολογιών. Από ό,τι άκουσα είχαμε κοινέ θέσεις, έχουμε κοινού στόχου. Λοιπόν, με τη δουλειά μας και την προσπάθειά μας θα καταλήξουμε σίγουρα σε χρήσιμες λύσεις και κοινέ λύσεις. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω, όπως ανέφερε και η συγκητής, ότι η προθεσμία της τροπολογίας είναι η 11 Οκτωβρίου, 12 μεσημέρι, ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 8 Νοεμβρίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών στις 5 Δεκεμβρίου. Πάμε στο επόμενο σημείο. Στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Ντάνκεν είναι ο μας. Και θα αρχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων. Όσον αφορά τις τροπολογίες των συναδέρφων σχετικά με το σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και θα ακούσουμε τον εισηγητή πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ να ακούσω τα σχόλια, αλλά εξαιτία των ε, διαδηλώσεων θα πρέπει να φύγω γρήγορα. Ε, δεν θέλω λοιπόν να μακρηγορήσω, προτιμώ να ακούσω τους συναδέρφους. Καλώς. Αρχίζουμε τότε με τους σκιώδεις εισηγητές. Τον κύριο Μπέλετ τον είχα δει εδώ, αλλά Τώρα δεν το βλέπω. Θα δώσω τότε το λόγο στην κυρία Νταλή που αντικαθιστά την κυρία Κούντραν. Παρακαλώ, Μίριαμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Τάνκεν, και για το χρόνο που κερδίζουμε. Αντικαθιστώ λοιπόν την κυρία Γκούτελαντ, η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Καταλαβαίνω και από εκείνη ότι οι διαπραγματεύσει ανάμεσα στον εισηγητή και τους οι εισηγητές προχωρούν θετικά και επικοδομητικά. Και γι' αυτό θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Θα σας παρουσιάσω ποια είναι η δικιά μας η θέση των σοσιαλιστών. Λοιπόν, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ένα σωστό σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών είναι ζωτική σημασία. Πιστεύω ότι μετά από τη Συμφωνία των Παρισίων είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί στο δρόμο για το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα υπέρ των κοινωνιών μας. Και η δικιά μας η ομάδα θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη φορά πρέπει να τα καταφέρουμε. Η ομάδα μας θέλει το σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών να είναι αυτό που πάντα θέλουμε να είναι ένα προοδευτικό σύστημα το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών με βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, σταθερό σύστημα το οποίο να προσφέρει σταθερότητα και στις επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να επενδύουν σε τεχνολογίες ε, καθαρής ενέργειας. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Το πρώτο που πρέπει να γίνει, το σύστημα επιστώσεων εκπομπών έχει παραμείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε ισχύ και πιστεύω ότι δίνει ένα στραβό μήνυμα. Η μεταρρύθμιση που διαπραγματευόμαστε είναι μια ευκαιρία που πρέπει να δράξει η Ευρώπη προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση και να πετύχει τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της σύντομα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς υποβάλλουμε διάφορες τροπολογίες οι οποίες οδηγούν σε περισσότερες μειώσεις των εκπομπών βάσει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι σαφές ότι πρέπει η γραμμική μείωση να αυξηθεί για να μην υπάρξουν περισσότερες, περισσότερη διάθεση δικαιωμάτων στην αγορά. Επίσης, χαιρόμαστε που το σύστημα θα βάλει ένα όριο στην ε, ε, δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων και θα ελέγξει καλύτερα το σύστημα πληστοριασμών. Η δωρεάν ε, διάθεση δικαιωμάτων πρέπει μόνο κατά εξαίρεση και για περιορισμένο χρονικό διάστημα να γίνεται. Συμφωνούμε λοιπόν για το 5% όσον αφορά τους πληστοριασμούς, αλλά πρέπει να μειωθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον πρέπει τα έσοδα επίσης από τους πληστηριασμούς όσον αφορά ε, τις, ε, τα δικαιώματα εκπομπών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβαλλοντικούς και μόνο στόχους. Το σύστημα πρέπει να είναι επίσης δίκαιο, πρέπει να είναι περισσότερο ακριβές το σύστημα διάθεσης δικαιωμάτων, να δίνεται μόνο όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα, μεταφοράς επιχειρήσεων δηλαδή αλλού, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Η συνεχής ενημέρωση επίσης των κριτηρίων είναι σημαντικό, έτσι ώστε η καινοτομία να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του συστήματος με τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα. Στηρίζουμε επίσης και την ενημέρωση των επιπέδων παραγωγής, έτσι ώστε η αγορά να είναι πιο δυναμική. Πιστεύουμε ότι προκειμένου το σύστημα να είναι πιο δίκαιο, πρέπει να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια κεντρική διαχείριση που να έχει να κάνει και με τις τιμές ηλεκτρισμού. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να στηρίζουν και άλλοι να μην στηρίζουν το σύστημα. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Κάτι άλλο πολύ βασικό για μας είναι αλληλεγγύη. Κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω σε αυτήν την ε, μεταβίβαση σε μια κοινωνία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις κοινωνικές πτυχές. Το και προτείνουμε ένα νέο μεταβατικό ταμείο το οποίο θα στηρίξει τα μέτρα ε, αυτά που θα χρειαστούν για την μεταβίβαση στην κοινωνία χαμηλού άνθρακα. Πιο αργά να μιλάτε, πιο αργά να μιλάτε, γιατί μιλάτε υπερβολικά γρήγορα, διαβάζετε γρήγορα. Το σύστημα αυτό λοιπόν πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα στο μέλλον και γι' αυτό προτείνουμε να ενισχύσουμε το Ταμείο Κοινοτομίας. Χρειάζεται έρευνα και επενδύσεις που θα στηρίξουν και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, είμαστε πεπισμένοι ότι το σύστημα αυτό μπορεί να λειτουργήσει καλά, να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο για να έχουμε μείωση της, το άνθρακα αλλά και περισσότερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη και καινοτομία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα και από μένα σε όλους. Έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις όσον αφορά τα βασικά ζητήματα του φακέλου αυτού. Ο συντελεστής πρώτα απ' όλα γραμμικής μείωσης. Είναι σαφές. Εμείς ως ΕΛΚ το στηρίζουμε. και το 2,2% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας βρίσκει σύμφωνους γιατί πρόκειται για μια φιλόδοξη πρόταση. Έχει να κάνει με τους δείκτες με τους οποίους συμφωνήσαμε με μάλλον τα εθνικά, τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές στο INCD που συμφωνήσαμε στο Παρίσι. Το στηρίζουμε και οι διεθνείς εταίροι. Τώρα, όσον αφορά το auction share, που αποτελεί επίσης τους πληστηριασμούς δηλαδή που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της πρότασης. Δεν θέλουν 57%, 52%. Γνωρίζουμε ότι πολλοί φορείς μιλούν για την απόφαση του Συμβουλίου του 2014, που φυσικά και σεβόμαστε. Και το Συμβούλιο, μάλλον υπενθυμίζω εδώ, ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου λένε ότι το μερίδιο δικαιωμάτων σε πληστηριασμό δεν πρέπει να μειωθεί. Δεν αναφέρεται ποσοστό, οπότε εμεί δεν αφισβητούμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, καθόλου. Αλλά ο υπολογισμός μας ξεκινάει από τη δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων από την αρχή της τρίτης περίοδου. Γι' αυτό και καταλήγουμε εμείς στο 52% αντί για το 57%. Κάτι το οποίο θα δώσει περισσότερο περιθώριο ελιγμών για διάθεση δωρεάν δικαιωμάτων. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν δίνουμε δωρεάν δικαιώματα σε όλους, αλλά μόνο σε επίπεδο 10% για την καλύτερη επίδοση των εγκαταστάσεων. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει κίνητρο για παρετέρω μείωση των εκπομπών διεξουδίου του άνθρακα στο μέλλον. Όσον αφορά τώρα το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για την αυτιλία, την αεροπορία κτλ. Νομίζω ότι για τους δύο αυτούς τομείς υπάρχει συνένεση εδώ ότι πρέπει να γίνει περισσότερη προσπάθεια για να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με άλλους τομείς του συστήματος. Η διάθεση δικαιωμάτων λοιπόν αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της πρότασης. Έρχομαι τώρα στα θέματα της ε, ανάλυσης της αγοράς. Τόμους που νομίζω ότι όλοι εδώ πέρα σέβονται λέει ότι η σημερινή πρόταση που προτείνουν διάφορες ομάδες λέει ότι η πρόταση αυτή για το τέταρτο στάδιο θα οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη για κάποιους μεγάλους τομείς. Το το βιομηχανία για παράδειγμα. Ναι, ο κύριος Σίχαρ θα έρθει αργότερα, απαντάει σε παρατήρηση εκτός μικροφώνου ο κύριος Μπέλετ. Θα έρθει σίγουρα. Λοιπόν, παραθέτω, συνεχίζω να παραθέτω τι άλλο λέει ο Βόιτεξ. Που και οι πράσινοι φίλοι μας σέβονται. Λέει λοιπόν ότι το στάδιο αυτό 4, μια τέτοια πρόταση, θα οδηγήσει σε μεγάλα κέρδη για μεγάλους τομείς, ενώ άλλοι τομείς όπως η βιομηχανία και άλλοι μπορεί να δουν τα κέρδη τους να μειώνονται και να πληγεί και η ανταγωνιστικότητά τους. Πολύ περίεργο λοιπόν που φαίνεται να καταστρέφονται κάποιοι τομείς από την πρόταση αυτή. Αυτή η σε επίπεδα προσέγγιση λοιπόν μπορεί να είναι και καταστροφική. Έρχομαι τώρα στα κριτήρια. Προτείνουμε να έχουμε φιλόδοξα κριτήρια, benchmarks, αλλά να καθοριστούν πριν την αρχή της νέας περίοδου εμπορίας, για να υπάρξει μια λογική πορεία στο υπόλοιπο του συστήματος, στην υπόλοιπη διάρκεια. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι υπάρχει σταθερότητα, προβλεψιμότητα και λογικά κριτήρια μέχρι το τέλος της περίοδου που να βασίζονται στην πραγματική επίδοση. Και όχι να προβλέπουμε για το 2020-2030 για στοιχεία που έχουμε από το 2008. Θα ήταν εντελώς παράλογο κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα την ποιοτική αξιολόγηση, Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ότι πρέπει να γίνεται αυτή η ποιοτική αξιολόγηση. Ελπίζω να βρούμε τα σωστά κριτήρια και να στηρίξουμε όλες οι πολιτικές ομάδες να μην καταργηθεί αυτή η ποιοτική αξιολόγηση. Το CSCF που πρόκειται για τον διατομιακό διορθωτικό συντελεστή είναι κάτι που στηρίζουν επίσης πολλές ομάδες. Το είπατε κι εσείς. Είναι καλό που και οι σοσιαλιστές είναι υπέρ της αρχής αυτής. Συνεπώς την στηρίζουμε αυτή την αρχή. Αναφερθήκατε σε μια δυναμική διάθεση δικαιωμάτων που επίσης στηρίζουμε. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο και πτυχή, Πρόεδρε, είναι, τα, ε, είναι το έμεσο κόστος. μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στήριξη για μια εναρμονισμένη προσέγγιση μέχρι κάποιο επίπεδο, όχι μόνο στην ομάδα μας, αλλά και σε άλλες πολιτικές ομάδες ισχύει. Πολύ θετικό αυτό. Αλλά υπάρχει πλήρης αντιστάθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μια δυσκολία παραπάνω. Πρέπει να δούμε κατά πόσο χώρες μέλη μπορούν να δώσουν περισσότερη στήριξη από το εθνικό επίπεδο και να υπάρξει έτσι μια, ένα συνδυασμός της εναρμόνισης με την ευελιξία του εθνικού επίπεδου και έτσι να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι καλό που υπάρχει ενδιαφέρον και ανησυχία για αυτές που συμμεριζόμαστε όλες οι πολιτικές ομάδες. Και το τελευταίο μου, Πρόεδρε, είναι το εξή. Η... Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το σύστημα και οι συνέπειές του σε συνδυασμό με εθνικές πολιτικές, ενεργειακή ε, και τα κτλ. Πρέπει να έχουν τον ίδιο στόχο, την μείωση της ρήπανσης και πρέπει να εξετάσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες όλων αυτών των πολιτικών. Μερικές φορές πρόκειται για επικάλυψη στόχων, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό και να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους. Αυτές είναι οι κυρίες παρατηρήσεις μου όσον αφορά την πρόταση που εξετάζουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε τη δυνατότητα στον κύριο Εκχάουτ να εξηγήσει την θέση του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα βήμα προς τα πίσω. Ας πούμε πέρσι στο Παρίσι, όπου όλες οι πολιτικές ομάδες είχαν εκφράσει την ικανοποίησή τους, με ενθουσιασμό μάλιστα, για την επιτυχία που σημειώθηκε εκεί. Και όλες οι πολιτικές ομάδες τώρα αγωνίζονται για να πιέσουν τις χώρες μέλη να κυρώσουν αύριο κιόλας. Διότι φαίνεται πως είναι τόσο ουσιώδη όλα αυτά για μας. Έχετε δει τι έχουμε συμφωνήσει στο Παρίσι ή απλώς ήταν συμπαθητικό να βρεθούμε εκεί και να δίνουμε το χέρι ένα στον άλλο. Νομίζω ότι ε, το ότι είναι καινή η αίθουσα τώρα, λίγο πολύ, λέει πολλά πράγματα. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην ε, πολιτική περιβάλλοντος. Και η Επιτροπή ΕΝΒΗ, η Περιβαλλοντική Επιτροπή, είναι το πιο σημαντικό μας εργαλείο. Και δέστε την αίθουσα. Δεν υπάρχουν σχεδόν, σχεδόν ευρωβουλευτές. διότι οι περισσότεροι έχουν παραιτηθεί. Αυτό συμβαίνει εδώ. Άρα, από τα πιο σημαντικά εργαλεία που διαθέτουμε για να κάνουμε κάτι για να εφαρμοστεί η Συμφωνία του Παρισιού, δέστε τι πολιτική υποστήριξη βρίσκει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που έχω. Και πριν αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες, με βαλώματα στο σημερινό σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί, ας εξετάσουμε γιατί υπάρχει το πρόβλημα αυτό, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον. Δεν μπόρεσα λοιπόν να δαγκώσω τη γλώσσα μου και να μην κάνω την ε, κοινική παρατήρηση στον κύριο Μπέλετ που λέει για Thomson Reuters και ρίχνει τόσο φως μήπως να μελετήσει όλες τις μελέτες τους που λένε ότι το τρέχον σύστημα δεν λειτουργεί και χρειάζεται εκ νέων, ε, συγγνώμη, εκ βάθους αναδιάθρωση και δεν υπάρχει τέτοια πρόταση τώρα. Λέμε, να εδώ ε, λίγο carbon leakage εκεί, κάτι άλλο. Δεν λένε αυτά οι μελέτες Thomson Reuters. Λένε για υπερπροσφορά του συστήματος αυτού 2,5 δις μέχρι το 2020 πιστοποιητικών. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Και εδώ εμείς μιλούμε για ελάσσονα θέματα. Και να σας εξηγήσω γιατί διαρωτώ με όλο και περισσότερο αν χρειάζεται πραγματικά να επενδύσω στην βελτίωση του συστήματος. Γιατί αν δείτε την παρούσα πρόταση, εάν δεν κάνουμε τίποτα για το σύστημα ETS, αν το αφήσουμε όπως είναι το σύστημα αυτό των ε, διοξιδίων. Θα σταματήσουν όλοι οι κανόνες για το carbon leakage μέχρι το 2020. Όλες οι εξαιρέσεις, το άρθρο 10Γ και όλα αυτά, θα σταματήσουν, θα πάψουν να ισχύουν το 2020. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Πολλοί ανησυχούν γιατί θα σταματήσουν οι κανόνες για το carbon leakage. Εγώ δεν ανησυχώ. Η μόνη βελτίωση που κάνει, που επιφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μόνο που κάνει, είναι να αυξάνει στο 2,2 τον συντελεστή γραμμικής μείωσης. Και αν δείτε τι σημαίνει αυτό για τη μείωση των πιστοποιητικών, θα δείτε ότι είναι περίπου 400 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Στην πρότασή της, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κερδίζει 400 εκατομμύρια πιστοποιητικών, allowances. Από τα 2,5 δισεκατομμύρια. Ταυτόχρονα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ευγούν από το MSR 250 ε, εκατομμύρια και να μπουν στο νέο αποθεματικό. Συνολικά 400 εκατομμύρια. Άρα 400 εκατομμύρια που κερδίζουμε τα παίρνει τώρα από την τρίτη φάση και το βάζει στην τέταρτη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι τελικό το κέρδος για το περιβάλλον από όλη αυτή την υπόθεση, τίποτε. Μπορούμε να καταψηφίσουμε τα πάντα τότε. Ίσως να μην φτάσουμε ούτε καν σε συμφωνία και δεν με πειράζει κιόλα, διότι δεν υπάρχει τελικό κέρδος για το περιβάλλον. Και αυτά, όταν συζητούμε την συνέχεια πρέπει να δοθεί στο Παρίσι, 5 ευρώ ανατόνο διοξιδίου του άνθρακος. Α, και ορισμένοι λένε ότι μπορεί να φτάσουν και στο 2,4 ο συντελεστής. Στην πραγματικότητα πρόκειται μονάχα για κερδοσκοπία. Έχουμε ένα, ένα, δυσλειτουργικό μηχανισμό, δεν υπάρχει κανένα κέρδος τελικός για το περιβάλλον και αυτά συζητούμε τώρα μετά το Παρίσι. Αν όντως αυτό συμβαίνει, τότε όπως ε, την άλλη φορά, ναι, την επόμενη φορά τότε ούτε την άλλη δεν βλέπω εδώ, ούτε την ΚΟΥΕ βλέπω εδώ, τότε και τι καθόμαστε και ασχολούμαστε. Αυτά διακυβεύονται και πρέπει να τα συζητήσουμε πολύ πιο ενεργά για να δούμε τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε πραγματικά το σύστημα και θα κάνουμε και κάτι για το πλεόνασμα των πιστοποιητικών. Και μπορούμε τότε να συζητήσουμε και το carbon leakage, αλλά πριν να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα λειτουργικό. Του χρόνου η Κίνα θα αρχίσει το εθνικό της πιλωτικό πρόγραμμα για το ETS και μετά από λίγα χρόνια θα αρχίσει να εμπορεύεται τα πιστοποιητικά. Αν μιλήσουμε μόνο για το carbon leakage, τότε ας δούμε και τι κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί αρχίσαμε να μιλούμε για το carbon leakage, διότι το κάνουμε αυτό εάν ο υπόλοιπος κόσμος δεν κάνει τίποτε. Όμως ο κόσμος κινείται ταχύτερα και εμείς καθόμαστε και συζητούμε τα χθεσινά. Και αυτό με λυπεί ιδιαίτερα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εύη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμερίζομαι πολλά από αυτά που είπε ο συνάδελφος Εκχάουτ. Κάθε παρέμβαση που έκανα μέχρι τώρα για το θέμα αυτό αποτελούσε απόπειρα περιγραφής των ελλείψεων που γνωρίζουμε πολλοί από εμά όσον αφορά αυτή την πολιτική. Όπως υπενθυμίστηκε αυτή η πολιτική είναι ένας πυλώνας ε, των πολιτικών της Ένωσης για το κλίμα. Ένας πυλώνα όμως δεν ε, στηρίζει τίποτα, δεν πετυχαίνει κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι οι μειώσεις των εκπομπών που διαπιστώσαμε ε, οφείλονται σε μικρέ παρεμβάσει ενεργειακή απόδοση στην παραγωγή περισσότερο παρά πραγματικές, σε πραγματικές επενδύσεις για πιο, καθαρή, ε, πιο καθαρές επιχειρήσεις. Η βούληση να κοιτάξουμε αλλού πρέπει να ξεκινήσει και το Κοινοβούλιο. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να κοιτάξουμε αλλού. Είναι προφανές και σαφές ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτή την πολιτική σήμερα ούτε αύριο αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε να ακολουθήσουμε μακροπρόθεσμη ανάλυση για λύσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, επί παραδείγματι, έχουμε τις έρευνες που πραγματοποιούνται σήμερα. Έρευνα της προστατικοποίησης του περιεχόμενου σε άνθρακα των προϊόντων. Άρα, να προσπαθήσουμε εν αυτή τη ενία να βρούμε μια λύση όσον αφορά τα προβλήματα από την αλλαγή του κλίματος. Στρεφόμενοι τώρα στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, συγκεκριμένο θέμα, θέλω να κράσω τις θέσεις μας όσον αφορά τους συμβιβασμούς που συζητούμε. Για μας η υψηλή τιμή του διοξιδίου του άνθρακος είναι η μόνη χρήσιμη προσπάθεια για να διαθεθούν χρήματα, να δοθούν χρήματα στα ταμεία των κρατών μελών που πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα για την ε, ε, ανάκαμψη και εξυγίανση των τομέων που καλύπτουν το σύστημα. Θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις δωρεάν άδειε ε, που δίδονται σε δημοπρασία χωρίς παρεκκλήσεις. Όσον αφορά τη γραμμική προσέγγιση, το 2,2 που αναφέρασα ποσοστό είναι πολύ χαμηλό και το 2,4 για μας είναι ένα βήμα πολύ μικρό. Και είναι πολύ δύσκολη βάση για να πραγματεύσουν το Συμβούλιο. Άρα πολύ αδύναμη αφετηρία. Πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Η πρόταση αυξήσεως το ρίο των 50.000 τόνων για την αυτοεξαίρεση των μικρών ε, επενδυτών είναι κάτι που μας βρίσκει αντιθέτους. Διότι έτσι θα επιτρέπαμε στους μικρούς ε, επιχειρηματίες να μην βάζουν, να μην εφαρμόζουν μέτρα αντιστάθμισης. Ανησυχούμε για την υποστήριξη στο ETS. Ίσως αυτό να ευνοήσει μόνο τις πετρελαϊκές εταιρείες που χειρίζονται τους σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου Brent. Και τα δηληστήρια θα μετατραπούν τελικά σε χώρους αποθήκευσης. Και είναι επικίνδυνο αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τα κράτη-μέλη για με τους χώρους αποθήκευσης του πετρελαίου αυτή είναι η θέση μας. Είμαστε αντίθετοι με τις συζητούμενες συμβαστικές λύσεις. Όσον αφορά αυτόν τον πυλώνα της πολιτικής του κλίματος, ε, η εικόνα μας είναι αυτή που είπα στην αρχή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για να αλλάξουμε κατεύθυνση. Αυτή είναι η βασική μας άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λίζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πρόταση που εξετάζουμε αποτελείται από ποικίλε πτυχές ε, και υπάρχει μια πολύ σημαντική πτυχή κατά την άποψη του ΕΛΚ, δηλαδή να... ένα θέμα που μας προβληματίζει. Υπάρχουν σήμερα βιομηχανίες που για λόγους τεχνικούς, λόγω τεχνικών δυνατοτήτων μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και είναι δυνατόν αυτές οι βιομηχανίες να μετακινηθούν τελικά, να πάνε αλλού. Είχαμε θετικές εξελίξεις στην Κίνα, ξέρουμε ότι η Συμφωνία των Παρισίων είναι πάρα πολύ καλή συμφωνία, αλλά όσον αφορά τα κίνητρα για τις ε, ανθρακοβόρες, ε, μάλλον ε, τις βιομηχανίες που παράγουν πολλές εκπομπές άνθρακα, είναι δύσκολο να βρούμε λύση διότι αντιμετωπίζουμε τους ανταγωνιστές που αντιμετωπίζουμε και στους κόλπους του ΕΛΚ πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες δωρεάν άδειε για ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως είναι χάλιβας, τσιμέντο, χημικά, λιπάσματα διότι αντικειμενικά αυτοί οι βιομηχανικοί τομείς θα πρέπει να θα αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω αυτής της προτάσεως και μάλιστα προβάλλουν και πολύ καλά επιχειρήματα για να δείξουν τα προβλήματά τους και αν ε, μόνο 10% των καλύτερων επιχειρήσεων παίρνουν τις ε, δωρεάν άδειε. Αυτή είναι η προτεραιότητα του ΕΛΚ. Θέλουμε περισσότερες δωρεάν άδειε και τη μείωση, των δημοπρασιών. Και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο ε, με αυτά που ακούω να λέγονται από κάποια κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένου και του κράτους μέλους που γνωρίζω καλύτερα που δυστυχώς δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί επίσημα. Ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες ε, θα υπάρξει μια γερμανική θέση που θα υποστηρίζει τις ιδέες. Η ιδέα είναι 1 ή 1,5% ε, βελτίωση όσον αφορά την ελεύθερη, τη δωρεάν ε, χορήγηση αδειών. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο. Το ΕΛΚ θα θέλει μια αύξηση του 5% και στο σύνολο. Άκουσα και τα όσα είπε ο Μπάς Αικχάουτ. Ασφαλώς μπορεί κανείς να ασκήσει και κριτική. Ας μην εντελώ όμως εντελώς ότι ε, καταργούμε τους μηχανισμούς CDM. Για να επιτύχουμε το 20% μείωση μέχρι το 2020, δυνατόν θα ήταν μόνο να χρησιμοποιηθούν και κονδύλια από τρίτες χώρες. Αυτό καταργείται. Αυτό είναι σωστό και το υποστηρίζουμε ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ας μην το λησμονούμε λοιπόν, άλλωστε και ο ΙΚΑΟ συζητεί στο Μοντρεάλ και είναι το μόνο που θα δεχόταν να αγοράζει δηλαδή ο μέσο των αέριων μεταφορών CDM και εμείς το καταργούμε αυτό. Και για να πάμε μέχρι το 2030 άλλα 20% κάτω χωρίς CDM νομίζω ότι είναι αρκετά φιλόδοξο. Ακούω επίσης Παρ' όλα αυτά, πολλοί, όχι μόνο μη κρατικέ οργανώσει, μη κρατικές οργανώσεις, αλλά και ε, κατασκευαστές ε, σταθμών παραγωγής που θα ήθελαν, ε, που φτιάχνουν εργοστάσια τα οποία θέλουν να μειώσουν εκεί την παραγωγή των οξυδίων του άνθρακα, ζητούν και εκεί πιο φιλόδοξους στόχους, όμως μόνο εφόσον εξασφαλίζεται η ασφάλεια σχεδιασμού για την ενεργοβόρο βιομηχανία. Έχουμε λοιπόν μια αγορά που είναι διχασμένη, καθώς και η βάση συμφερόντων είναι διχασμένη και πρέπει λοιπόν να λεφθούν υπόψη αυτά περισσότερο. Έχω τώρα και τις τροπολογίες 193 και 194 και ορισμένες άλλες σχετικά με τις εναερίες μεταφορές. Τις υποστηρίζουμε και χαίρομαι που ο συντονιστής Βιμ Φαντεκάμπ στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος τα υποστηρίζει. Αυτά εντός Ευρώπης. Θα δούμε όμως και τι θα κάνει ο ΕΚΑΟ εκτός Ευρώπης την επόμενη εβδομάδα. Θέλουμε προσέγγιση μέσα στην Ευρώπη. Δεν βρίσκω να είναι σωστό να επιβάλλουμε στη χαλιβουργία συντελεστή μείωση 0,43% και για την ενέργεια βιομηχανία μείωση της τάξης του 5%. Εάν δεν μπουν περισσότερες πιο φιλόδοξη στόχη. Άρα, μεγαλύτερη πίεση στον ε, τομέα των αέριων μεταφορών, κάπως όμως πρέπει να προσεγγίσουν οι στόχοι. Και αυτό είναι σημαντικό και διότι και άλλοι φορείς μεταφορών, όπως ο σιδηρόδρομος, που ασφαλώς είναι φιλικότερος στο περιβάλλον, χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα, είναι μέσα στο πλαίσιο του 43% του, της μείωσης. Μήπως πρέπει να ενισχύσουμε λίγο στο πλαίσιο αυτό τον φιλικό φορέα μεταφορών σιδηρόδρομο. Ας πούμε ότι βγάζει κανείς ένα εισιτήριο από Βρυξέλλες προς Φραγκφούρτη. Μπορεί να πετάξει κανείς με 15% συν 5% ή αν μπει στο τρένο Εκεί 100% ETS με μείωση 43% και με 100% δημοπράτηση. Χρειάζεται λοιπόν κάποια, να δοθεί κάποια άλλη κατεύθυνση, χρειάζεται και περισσότερη δικαιοσύνη. Τώρα μαζί με τον πρόεδρο, γνωρίζω ότι ο Ματίας Γκρότε έχει καταθέσει και αυτός παρόμοια τροπολογία, προτείνουμε να ενισχυθεί το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Χρειαζόμαστε δηλαδή περισσότερα χρήματα για να μπορέσει η κεντρική και ανατολική Ευρώπη να χτίσει σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Για αυτά να βασιστούμε στο άρθρο 10 γάμε, 10C. Εξακολουθεί να προβλέπεται στη, στην πρόταση της Κομισιόν η δωρεάν χορήγηση πιστοποιητικών Καταρχήν το έχουμε σταματήσει αυτό, όμως για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο κεντρική, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, σωστό είναι να ενισχυθεί το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Γιατί θα έχουμε τότε στα χέρια μας ένα μηχανισμό που επιτρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον, να δαπανίσουμε χρήματα δηλαδή για την ενίσχυση επενδύσεων στραμμένων στο μέλλον. Θα χαρώ πολύ αν μπορέσουν οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν την τροπολογία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βυσνιεύσκα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, από την αρχή να προβώ σε δύο γενικά σχόλια. Υπευλήθησαν κάποιες τροπολογίες στην έκθεση Duncan σχετικά με το σύστημα ETS Πολλέ τροπολογίε υπευλήθησαν γιατί το σύστημα πιστεύουμε δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει, κυρίω όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών. Εκφράσαμε αμφιβολίε για την προσέγγιση. Θα πρέπει να πετύχουμε του ίδιου στόχου με διαφορετικού τρόπου που είναι λιγότερο επαχθής από πλευράς φορολογικής και διοικητικής. Για κάποιο λόγο όμως αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια περιπλοκότατη μέθοδο. Θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη βεβαιότητας για τους τομείς που καλύπτονται από το ETS. Οικονομικούς τομείς, γενικά τον οικονομικό τομέα, αλλά και για ενεργοβόρες βιομηχανίες. Οι περισσότεροι από εμά βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα να επιβάλλουμε μεγάλο άχθος στους διάφορους τομείς, κάτι που θα έχει οικονομικό αντίκτυπο και υποφείλει στο σύστημα ETS. Κανείς δεν έχει σαφή εικόνα όμως, κάποια ιδέα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεύτερον, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις που θα προταθούν. Αυτό που έχουμε εδώ για την ώρα αυξάνει το χάος και την αβεβαιότητα για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο μηχανισμό ETS. Υπάρχει μια μετακίνηση προς δημοπράτηση και προς την χορήγηση ελευθέρων αδειών προς κάποιες βιομηχανίες. Υπάρχουν διάφορες λύσεις για τα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τη διάρθρωση των τιμών των αδειών που θα σχετίζονται με οικονομική ανάπτυξη ενδεχομένω, αλλά επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα. Κάποιοι από εμά ίσως θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθούμε τις βιομηχανίες που είναι πολύ σημαντικές, μονάδες παραγωγής ενέργειας ε, στις περιοχές μας και στις περιφέρειές μας. Αλλά μια τέτοια προσέγγιση θα οδηγούσε σε προβλήματα. Θέλουμε πιο ισορροπημένη λύση, πιο βιώσιμη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με διαρροή άνθρακα. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, κάποιες πιο μεγάλες, πιο προβληματικές. Υπάρχουν προτάσεις των πρασίνων και των σοσιαλιστών Εάν ακολουθήσουμε τις δικές τους λύσεις θα οδηγηθούμε σε μεγάλη αβεβαιότητα για προστατευμένους τομείς που παρέχουν ε, θέρμανση. Θα πρέπει να μετακινηθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος εκτός ε, του τομέα του ETS. Το θέμα είναι να μην χάσουμε τα πάντα με τις προτείνομενες λύσεις. Το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές Θέλω να εξαιρεθεί το 10% των καλύτερων μαθητών του τομέα. Και βέβαια έχουμε και διατομιακό διορθωτικό παράγοντα που προτείνεται. Εάν πάρουμε 10% των μονάδων που δεν παίρνουν αρκετές άδειε, αρκετά ποσοστά, θα είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουν. Και θα υποφέρουν διπλά. Πρώτα απ' όλα δεν θα πάρουν τις ελεύθερες άδειες, τις δωρεάν άδειες, διότι αυτό εξαρτάται από το επίπεδο των εκπομπών, αλλά θα εξαιρεθούν και από άλλο στάδιο εφαρμογής του μηχανισμού. Και αυτό θα ήταν απειλή για τις εταιρείε για τις επιχειρήσεις που ηγούνται στον τομέα. Αυτό θα επηρεάσει την καινοτομία και η καινοτομία υποτίθεται ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους της νομοθεσίας για το ETS. Μέχρι τώρα είδαμε οι πιο ε, καινοτόμες μονάδες να μην συμπεριλαμβάνονται στο 5% των αποτελεσματικότερων μονάδων. Προφανώς εξαρτάται και από την όλη υποδομή τους. Για αυτούς τους λόγους, στις τροπολογίες που υπέβαλα, προτείνω να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τη βάση ούτως ώστε να μιλάμε για το 20% των αποτελεσματικότερων μονάδων και η αξιολόγηση να γίνεται βάσει των πλέον προσφάτων στοιχείων και πληροφοριών. Για να είμαστε δίκαιοι. Περιγράφω τις ιδέες αυτές τροπολογίσμου τροπολογίες μου και προσπαθώ να καλύψω τα διάφορα ζητήματα που σας παρουσίασα στις τροπολογίες μου. Προφανώς θα πρέπει να δούμε τι προτάθηκε στο Συμβούλιο το 2014 και προτείνω να δούμε και τις εκπομπές των βιομηχανικών διαδικασιών που εκεί ίσως να υπάρχουν και κάποια προβλήματα για τη μείωση των εκπομπών και το ρόλο των δασών πρέπει να εξετάσουμε, τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα δάση. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός. Μετά έχουμε το Ταμείο Ξυγχρονισμού. για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν οι φτωχότερες χώρες. Πιστεύω ότι το Ταμείο Ξυγχρονισμού θα πρέπει να παραμείνει και πρέπει να στηρίξουμε τους δικαιούχους του Ταμείου. Τώρα για την εναρμόνιση του συστήματος αποζημιώσεως για το έμεσο κόστος Υπάρχει διαφορά δυσκολιών που αντιμετωπίζουν διάφορες χώρες για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς στόχους του ενεργειακού τομέα και πρέπει να υπάρχει μια αντιστάθμιση των προβλημάτων. Υπάρχει και η ενεργειακή φτώχεια ε, που θα πρέπει να μην τη λησμονούμε και θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτό το πρόβλημα. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κ. Φαρέ πρέπει να φύγει μετά την ψηφοφορία. Ζητάει συγγνώμη. Έπρεπε να πάει στη Μαδέρα σε μια σημαντική συνεδρία. οπότε μου έδωσε τι παρατηρήσεις του σχετικά με τις τροπολογίες που έχει ο ίδιο υποβάλει. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις του λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, ότι είναι ο μόνος ε, στόχος η ναυσιπλοεία που δεν συμμετέχει στους στόχους. Ότι υπάρχει αύξηση 44% μέχρι το 2030 και 60% σε σχέση με το 2050 αν συγκρίνουμε με την εποχή της δεκαετίας του 90. 30,7% των εκπομπών μέχρι το 2050, το 2050 θα έχουν αυξηθεί πολύ αν δεν υπάρξει καμία παρετέρω ρύθμιση. Η αύξηση αυτή των εκπομπών προφανώς και είναι σύμβατη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση μέχρι το 2030, επειδή υπάρχουν και στόχοι των Παρισίων. Ο κύριος Φαρία προτείνει ένα ουδέτερο ταμείο για το κλίμα, το οποίο θα βοηθήσει να επιτεθούν οι στόχοι του 2030 και να ευθυγραμμιστούμε με τους στόχους των Παρισίων. Να μιλάτε πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει το σημερινό σύστημα ελέγχου βέβαια των εκπομπών. Πρέπει να υπάρχει συνδυασμό με αυτό για να παραμείνει όσο γίνεται πιο χαμηλό το κόστος για τους πλειοκτήτες και τις αρχές. Θα λειτουργήσει ω εκ, ε, ως εξής. Οι πλειοκτήτες οι οποίοι φτάνουν ή φεύγουν από ευρωπαϊκούς λιμένες θα πρέπει ή να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών για να καλύψουν τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα ή να πληρώνουν ένα ισοδύναμο ποσό στο ταμείο το οποίο συλλογικά θα φροντίζει για την ε, κατανομή δικαιωμάτων και έτσι θα μειωθούν αυτά ε, στο ίμιση. 20% των εισοδημάτων από τα δικαιώματα θα επανεπανδύονται προκειμένου τα σκάφη και ευρωπαϊκό στόλος να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Έτσι πιστεύουμε ότι στηρίζεται και η μείωση του διεξουδίου του άνθρακα και η καινοτομία. Περίπου ένα δισεκατομμύριο θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε κυρία Καρντίνη τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω να επικεντρωθώ επί μιας προτεραιότητας που θεωρώ ότι είναι σημαντική, το έμεσο κόστος. Πρέπει να εξαλείψουμε τις τρευλώσεις που δημιουργούνται στο σύστημα ETS, που δημιουργεί εσωτερικό dumping. Όταν η υποζημίωση του έμεσου κόστους γίνεται επιθελοντικής βάσης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ελάχιστα κράτη που εφαρμόζουν αυτό το μέτρο, διότι υπάρχουν και ελάχιστα τα κράτη που μπορούν να το κάνουν. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα που έχουν τα κράτη να αποζημιώσουν εθελοντικά, ε, θα ήταν απλές κρατικές ενισχύσεις. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να μείνει όσο έχει. Και δεν καταλαβαίνω τις αντιστάσεις που υπάρχουν από ό,τι ακούγονται στους διαδρόμους υπάρχουν αντιρρήσεις από κάποια κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε να καταργήσουμε το μηχανισμό των αποζημιώσεων. Θέλουμε απλώς ο μηχανισμός να είναι ισότιμος για όλους. Το πρόβλημα αυτό εξάλλου θα γίνει όλο και πιο σοβαρό, πιο σημαντικό και θα αυξήσει με δραματικό τρόπο τις διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα υπάρχει διαφορά στην ανταγωνιστικότητα διαφόρων επιχειρήσεων ανάλογο με την έδρα του στα διάφορα κράτη-μέλη. Κάτι που θα γίνει δραματικό. Αν παραμείνει αυτό το, αυτή η καθεστική ατάξη και αν από τη 2021-2030 με τα μέτρα που λαμβάνουμε θα έχουμε ε, δικαιώματα ETS που θα κοστίζουν μεταξύ 25 και 40 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι σε ελάχιστα χρόνια το μειονέκτημα, το ανταγωνιστικό των επιχειρήσεων που κινούνται σε χώρε που δεν έχουν εθνική αποζημίωση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα είναι σε πολύ μειοντική θέση. Αρκετά άτομα εντό του Κοινοβουλίου ε, ασχολούνται με το θέμα, το θεωρούν σημαντικό. Πάνω από 70 τροπολογίες είδαμε πάνω σε αυτό. Επέρα των ε, τροπολογιών Ήτρε και Ένβη. Ε, θα ζητούσα λοιπόν από το Κοινοβουλίο και από τους συναδέλφους να παρακολουθούν προσεκτικά πώς προχωράει το πράγμα Ευχαριστώ τους εισηγητές μας που προωθούν το θέμα αυτό. Όμως πιστεύω ότι πρέπει πραγματικά και πάνω σε αυτό να είμαστε φιλόδοξοι. Οι προτάσεις είναι πολλές και διαφορετικές. Αυτό που προτείναμε εμείς θεωρούμε σαν τελική αντιπροσωπεία ότι κάναμε κάποιες προτάσεις που θεωρώ ότι η πρότασή μα είναι σημαντική, ε, συγκεκριμένη μάλλον. Να δημιουργήσουμε σύστημα αποζημιώσεων, αντισταθμίσεων που θα δημιουργείται από τα έσοδα μιας ποσότητας χ από, όλε τις, από τα δικαιώματα που θα δημιουργηθούνται ανάμεσα στο 2021 και 2030. Αυτό αναφέρει στην τροπολογία μα 381. Θα πρέπει όμως παρόλα αυτά, αν δεν βρούμε αυτή τη λύση, να βρούμε ένα άλλο σύστημα. Να δημιουργήσουμε τη βάση Ίσως χωρί να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δει α, τις λεπτομέρειες. Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Θα πρέπει όμως να θέσουμε τη βάση για ένα σύστημα που θα καθιστά πραγματικά εναρμονισμένο το σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να υπάρχουν ίσες, ίσα δικαιώματα. Το θέμα των αντισταθμίσεων που δίνουν στις επιχειρήσεις να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη ισότιμα. Δεν έχουμε μόνο το άμεσο κόστος, αλλά και το έμεσο. Και δεν κατανοώ πώς μπορούμε να σκεφτούμε ότι δεν θα έχουμε έναν μηχανισμό αποτελεσματικό σε αυτόν τον τομέα. Διότι, επαναλαμβάνω, στο μέλλον με τις αλλαγές που θα κάνουμε, με τα πιστοποιητικά που θα κοστίζουν πιο πολύ για να λειτουργεί το σύστημα, εάν παραμείνουμε έτσι θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες διαφορές. Στην τροπολογία μας δεν αναφέρουμε ακριβώς τα ποσοστά. Αναφέρθηκε ένα 3%. Ένα 3% θα ήταν ανεπαρκέστατο, το ξέρουμε. Ας αφήσουμε στην Επιτροπή να αποφασίσει την αξιολόγηση των ποσοτήτων. Ποιο είναι το απαραίτητο ποσοστό για να δημιουργηθεί ένα πραγματικό σύστημα εναρμονισμένο για όλη την Ευρώπη. Όμως πιστεύω ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα. Και είμαι βαθιά πεπισμένη επίσης ότι θα πρέπει, και αυτή είναι η δεύτερη μου προτεραιότητα, ότι θα πρέπει, λέγω, να δώσουμε προσοχή στο επίπεδο των δωρεάν δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν στη βιομηχανία. Να μην πηγαίνουν ε, στις βιομηχανίες που ρηπαίνουν, αλλά στις καλύτερες βιομηχανίες, εκείνες που σέβονται όλες τις ε, απαιτήσεις που έχουμε θέσει και θα εξακολουθούμε να θέτουμε ε, όσον αφορά το θέμα, που έχουν τι καλύτερε επιδόσει. Μόνο σε αυτέ πρέπει να πηγαίνουν. Θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Διότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο πολύ γρήγορα αλλάζει κανεί δρόμο ε, και μπορούν να φύγουν οι βιομηχανίε. Βιομηχανία σημαίνει θέση απασχόληση. Θέση απασχόληση σημαίνει οι νέοι μπορούν να εργαστούν, οι οικογένειες που μπορούν να ζήσουν. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο Το ότι κάποιο δημιουργεί μια επιχείρηση, αλλά και η επιχείρηση δημιουργεί θέσει απασχόληση, παίζει κοινωνικό ρόλο. Πρέπει να βοηθούμε την βιομηχανία να πηγαίνει καλύτερα, αλλά μην την πιέζουμε αρκετά και να μετεγκατασταθεί, διότι θα δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα με τη μετεγκατάσταση. Θα δημιουργήσουμε ζημίε. Λοιπόν, έμεσο κόστο και τι δωρεάν ποσοστώσεις που θα δίδονται στι ε, καλύτερε βιομηχανίε που έχουν καλύτερε επιδόσει. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπάλτζο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ συζητούμε για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν δύο ακραίε θέσεις. Η μία, η πρώτη, δεν την πολύ ακούμε εδώ, την ακούμε από τη βιομηχανία που λέει ότι το σύστημα αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο. Η άλλη άποψη είναι εκείνη των πράσινων ριζοσπαστικών που αυτό που θέλουν από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών είναι σιγά σιγά το τοπίο να αλλάξει, να μην υπάρχουν ορυκτά καύσιμα, γιατί σιγά σιγά το σύστημα αυτό θα αναγκάσει τις χώρες μέλη να αλλάξουν πορεία, να μετακινηθούν προς μια πράσινη αντιμετώπιση. Αυτό που είναι βέβαιο όμως και πρέπει εδώ να υποθεί είναι ότι το σύστημα αυτό καθε αυτό διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφώνεται με τις υποχρώσεις που έχει αναλάβει σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διεξουδίου του άνθρακα. Αυτό είναι σίγουρο. Και επίσης είναι σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καταφέρει περισσότερα για το 2030, όπου προβλέπουμε 40% μείωση των εκπομπών, αλλά Φανταστείτε ότι θα πάμε παραπάνω, όχι 50%, 60%. Πώς θα επιτευχθεί αυτό. Δεν θα πρέπει να επιτευχθεί με τον εξή τρόπο. Υπάρχει μια επιχείρηση στην Ουγγαρία με 10.000 υπαλλήλους. Μπορεί να μην είναι πολύ σύγχρονη η εταιρεία, αλλά αν μη όλο έχει προσπαθήσει να εξυγχρονιστεί. Όμως με τις καλύτερες επιδόσεις έχει τρία δικαιώματα και μετά αναγκάζεται να κλείσει. Δεν είναι το ίδιο όπως αν έχει κανείς ένα παλιό αυτοκίνητο και μετά το δίνει και αγοράζει ένα καινούριο για να προσπαθήσει ε, να βελτιώσει τις επιδόσεις στο περιβάλλον. Όχι, εδώ πέρα πρόκειται για το κλείσιμο μιας ολόκληρης επιχείρησης και πάνε στράφη προσπάθειες που έχει κάνει. Παρόλο λοιπόν που λειτουργεί κανονικά, αναγκάζεται να κλείσει. Στην Ουγγαρία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλιακή ή αιωλική ενέργεια αποκλειστικά. Οπότε η κυβέρνηση και επιχειρήσεις πρέπει να φροντίσουν να βοηθήσουν. Τι γίνεται λοιπόν, έχουμε φιλόδοξους στόχους. Όπως είπα, την ενέργεια τώρα θα την πάρουμε από την Ουκρανία. Και στην Ουγγαρία θα κλείσει αυτό το εργοστάσιο, αυτή η μονάδα. Θα πέσουν μεν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά θα αγοράζουμε η ηλεκτρική ενέργεια από την Ουκρανία. Αυτό θα οδηγήσει την Ουκρανία να εκπέμπει περισσότερο αέρια του θερμοκηπίου. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μειώσει τελικά τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο απλώ μεταφέρονται οι εκπομπές στην Ουκρανία ή στην Κίνα. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για την προστασία θέσεων απασχόλησης, δηλαδή για την διαρροή άνθρακα όπως λέγεται, δεν μπορούμε να πετύχουμε την μείωση εκπομπών διεξουδίου του άνθρακα συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό πιστεύω, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί για την μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, έχοντας και το στόχο του 40% όπως είπαμε, τότε πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν ε, βλέπω να έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο. Α, παρακαλώ, η Πιλάρ. Ευχαριστώ. Θέλω να επιμείνω σε αυτά που είπε η κυρία Καρτίνη. Ήμουνα στην Επιτροπή Γεωργίας, γι' αυτό άρχισα να έρθω εδώ. Θέλω να επιμείνω, λοιπόν, όσον αφορά τις συνομιλίες για το κόστος και να πω ότι η ρύθμιση αυτή θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα δωρεάν δικαιώματα και τις μειώσεις. 2,2% πρέπει να είναι το πολύ, όχι παραπάνω. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερες και αλλιώς ο σκιώδης εισηγητής μας τα είπε. Αυτά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά ακούσαμε. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να τα καλύψω όλα. Σίγουρα θα επανέλθουμε και με τις τροπολογίες. Θέλω να τη δράσω όμως σε τρία πράγματα βάσει της συζήτηση που παρακολούθησα. Πρώτον, πώς θα βρούμε το σωστό δρόμο να προχωρήσουμε και πώς θα υπάρχει μια καλή ισορροπία για να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά το περιβάλλον, αλλά μην έχουμε και διαρροή άνθρακα, δηλαδή να, μην έχουμε, να προστατεύσουμε και τις επιχειρήσεις μας. Οι ερευνητές, οι εμπειρογνώμονες τα παρακολουθούν όλα αυτά και μέχρι τώρα είμαστε επιτυχείς. Τώρα για το μέλλον πώς θα είμαστε επιτυχείς. Αναφερθήκατε σε πάρα πολλά, στα κριτήρια, το να αποφύγουμε, να ελαχιστοποιήσουμε τον διατομικό διορθωτικό συντελεστή πώς θα πρέπει να έχει η μελλοντική νομοθεσία και πώς θα ενισχύσουμε την βιομηχανική καινοτομία. Πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας ε, τις νέες τεχνολογίες και ρηπαίνοντα λιγότερο το περιβάλλον. Είναι θέμα ισορροπία λοιπόν και αυτό είναι κάτι που απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ταμείο Καινοτομία, για παράδειγμα. Κάτι συγκεκριμένο τώρα σε σχέση με αυτά που είπε ο Σκιώδης η εισηγητής από το ΕΛΚ που αναφέρθηκε στην ενημέρωση των κριτηρίων. Κάτι είπε για το 2008 ότι βασιζόμαστε μόνο σε αυτά τα δεδομένα. Κοιτάξτε, η πρόταση της Επιτροπής είναι να χρησιμοποιούνται και παλιά και νέα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι κι πρέπει να συλλέγονται τα νέα δεδομένα από τις διάφορες αρχές Οπότε χρησιμοποιούμε και τα δύο. Τα πάμε στην Κίνα ή και σε άλλα μέρη, διαπιστώσαμε ότι αυτοί μας ζηλεύουν που έχουμε τόσο πρόσφατες πληροφορίες από την βιομηχανία μας. Άλλοι δεν τα έχουν καθόλου. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και να μην τα βγάλουμε από την εικόνα. Κάποιος ανδιαφέρθη ε, και μίλησε για την προβλεψιμότητα. ακριβώ. Για να πετύχουμε λοιπόν στην καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα, τα χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία. Κάτι άλλο τώρα, πώς θα βοηθήσουμε τις χώρες στην Ανατολική Ευρώπη να εξυγχρονίσουν τον ενεργειακό του τομέα. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ήδη από το 2014 συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο στο μείωσης. Και δεν έγινε αυτό επειδή θέλησαν να κάνουν το χατήρι της μιας πλευράς της Ευρώπης και να παραβλέψουν την άλλη πλευρά της Ευρώπης. Όχι, είναι γιατί οι διάφορες εκθέσεις που γίνονται αξιολόγησης δείχνουν ότι οι προκλήσεις είναι τεράστιες και στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό το αντιλαμβάνονται και οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και οι εμπειρογνώμονες. Και εμείς ως ε, θεσμικά όργανα έχουμε μπροστά μας την πρόκληση να κάνουμε τις σωστές προτάσεις, να δούμε τι θα γίνει με τις εξαιρέσεις και πώς θα προχωρήσει το νέο Ταμείο Εξυγχρονισμού έτσι ώστε να υποφεληθεί ο ενεργειακός τομέας και να εξυγχρονιστεί και αυτός εκεί που χρειάζεται. Ένα άλλο στοιχείο που θα έπρεπε να έχουμε υπόψη μας είναι πώς θα υπάρξει μόχλευση ώστε οι επενδύσεις που γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα να αποδώσουν περισσότερο. Αν πετύχουμε σε αυτή τη μόχλευση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, τότε θα καταφέρουμε ακόμα περισσότερο και θα είναι προς όφελος των χωρών μελών. Και τρίτον, για τις παρατηρήσεις των πρασίνων. Πολλή συζήτηση γίνεται και την παρακολουθούμε και εμείς κατά πόσο είναι αρκετά ισχυρό το σύστημα. Αν ρωτήσετε, τα διαφερόμενα μέρη έχουν διαφορετικές απόψεις από αυτού. Οι αναλυτές επίσης έχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους και οι ερευνητές. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Είχαμε υπόψη μα ότι οι επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων είπαν ότι πρέπει να έχουμε μια καλά λειτουργούσα αγορά άνθρακα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο το οποίο μας καθοδήγησε και στην πρότασή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις τελευταίες συζητήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος είπε ότι είναι ανοιχτή στον προβληματισμό για το πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτό το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ε, εκπομπών. Είμαστε ανοιχτοί. Ακολουθούμε, παρακολουθούμε τις συζητήσεις και αυτή που έγινε εδώ. Δεν είμαστε κλειστοί καθόλου, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έτσι και αλλιώς πρέπει να ακολουθήσουμε τα συμπεράσματα των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων του 2014. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα, για τα συμπεράσματα, ο εισηγητής μας για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ όλους όσοι συμμετείχαν στην σημερινή συζήτηση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Okay. I... I'm going now to remember the time. Να υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 8 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ.